Où sont les explications de vote Good. Empezamos por el informe de la señora Stiller. Αρχίζουμε από τη λέξη κυρία Στάιλερ. Για ε, τις δομικές κατασκευές. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι σημαντικός τομέας ε, οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας και η βελτίωση των προδιαγραφών των Ευρωπαίων πολιτών δεν, μπορούν να, δεν μπορεί να μελεί ένα τόσο σημαντικό τομέα. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός για την ασφάλεια είναι ο δομικός τομέας ε, και ο εξυγχρονισμός του. Φυσικά όλοι θέλουμε να έχουμε κατασκευή με χαμηλό κόστος και των σπιτιών μας και των δημοσίων κτίριων. Με την έκθεση αυτή έχουμε άρση των φραγμών της αγοράς, απελευθέρωση της αγοράς και εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Τα ωφέλη ε, της πρωτοβουλίας αυτής ε, θα ευνοήσουν ολόκληρη την Ευρώπη και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ε, ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων στον δομικό κλάδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλινόφσκι. Ο κύριος Αντωνιώτης έχει το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ, συνάδελφοι, όσοι δεν έχετε ευεξήγηση ψήφου, να εξέρχεστε ησύχω τη αιθούση. Δεν ακούω και τίποτα, αλλά ε, ε, είναι σημαντική σημασία που αποδίδει η Ευρώπη στον τομέα αυτό. Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τα οποία αφορούν 12 εκατομμύρια ε, πολίτες που απασχολούνται σε αυτό το τομέα. Η έκθεση Σανδέλφου Στάινερ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να καταρρύψουμε τους εθνικούς φραγμούς, τους διοικητικούς και τους τεχνικούς που εμποδίζουν την εμπορευματοποίηση των προϊόντων στις κατασκευέ στην Ευρώπη. να προχωρήσουμε ε, σε, έναν, ε, σε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά σε αυτόν τον τομέα. Αναγνωρίζω βέβαια την αναφορά που γίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον οικοδομικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι είναι απαραίτητο να ανακυκλώνονται τα οικοδομικά υλικά. Αυτό είναι ένα θέμα καθοριστικής σημασίας, κυρίως στον αγώνα μας ε, για την κλιματική αλλαγή. Δράτουμε λοιπόν τις ευκαιρίες για να επιστήσω την προσοχή σας και για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών συσκευών. Λοιπόν, αυτά που λέει η συγκήτρια είναι χρήσιμα αλλά δεν αρκούν. Πρέπει λοιπόν να ε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα στο εγγύς μέλλον εκ νέου και να διασφαλίσουμε σε όσους απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών υψηλότερη προστασία. Έχουμε μια τραγωδία εργατικών ατυχημάτων και αυτό αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Ελπίζω λοιπόν με τη δουλειά μας να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση για αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Αντωνιώτση. Για ένα λεπτό το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Κάθριν Στάιλερ. Είναι πολύ καλή η έκθεσή της. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε εναρμόνιση των δομικών ε, υλικών. Θα έχουμε καλύτερες κατασκευές και ε, με υψηλότερη ποιότητα και προδιαγραφές. Έχει σημασία αυτό και για τον ανταγωνισμό, ο οποίος βέβαια δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι τα κτίρια πρέπει να είναι ασφαλή και για τους χρήστες, αλλά και για τους χτίστες. Οπότε ε, έχει σημασία να υπάρχει αυτή η εναρμόνιση, βοηθάει και το εμπόριο και το ε, την οικονομία και ε, γενικότερα την ε, πρακτική στον τομέα των κατασκευών για πολλές χώρες στην Ευρώπη γιατί υπάρχουν ακόμα χώρες που είναι κακής ποιότητας στα οικοδομικά υλικά οπότε χρειάζεται καλύτερη πρακτική, καλύτερα προϊόντα με καινοτομία στην Ευρώπη. Επίση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι δεν θα πρέπει να βλάπτουν την υγεία αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται και τα υλικά. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Στάιλερ, πολύ καλή έκθεσή τη. Και θέλω να τονίσω και πάλι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύνολο του κατασκευαστικού τομέα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα ήρθε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας στο Λονδίνο και μας είπε ότι θα πρέπει να πούμε ε, ε, στο μηχανισμό στήριξης για την ενίσχυση του ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι προβλήματα άλλων. Αν παραμείνουμε στη λογική και στο συνειρμό, τι λέει, δεν δουλεύει η ευρωπαϊκή κοινοποίηση, άρα ας την ενισχύσουμε, να έχουμε περισσότερη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ότι έχω μια βαρκούλα και εξοκύλει και γέρνει, βάλτε με καπετάνιο σε υπεροκειάνιο. Όποιο και να είναι το πρόβλημα, πάντα η απόφαση, η πρόταση που έρχεται είναι περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ότι η λύση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έγκυκε η ώρα όμως που δεν θα μπορούμε να ε, διαφέρουμε τόσο πολύ και να ε, απομακρυνόμαστε και από τις αγορές και από τους πολίτες ε, όσα ευχολόγια και αν χρησιμοποιούμε και σε Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι η επεξήγηση ψήφου σας δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το αντικείμενο της έκθεσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είστε ελεύθερος να αγορεύετε στο κοινοβούλιο. Έκθεση της κυρίας Τριφλέρ τώρα ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Μαστέλλα. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη που προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο και μιλάμε για πάνω από 40% της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Με την πολιτική της αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει πολύ συγκεκριμένα τη δέσμευσή της ε, για την προστασία ε, των τρίτων χωρών και των πολιτών που χρειάζονται αυτή την προστασία. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η συμφωνία που υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου ε, και την συνυπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Θα ήθελα λοιπόν να επενθυμίσω ότι με βάση αυτή τη συμφωνία υπάρχουν δεσμεύσει και για τα κρατημέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταγράψει μια όλο και μεγαλύτερη δέσμευση όσον αφορά την ανθρωπιστική χρήση. Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορεί να ε, μπορέσουν να γνωριστούν καλύτερα και να αρχίσουν ένα διάλογο για να μην τίθεται σε κίνδυνο ο ρόλος και οι ε, στόχοι. Βεβαίως ε, αυτά θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με όσα έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Μαστέλα. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Αντινόρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω ότι η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα της ε, συναδέλφου κυρίας ε, Στρίφλερ, την οποία και ευχαριστώ και συγχαίρω, είναι μια έκθεση η οποία αφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται αποτελεσματικότερα ε, για να δώσει μια συλλογική απάντηση στο θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο σε επίπεδο και πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η βοηθεία να φτάνει καλύτερα στους πολίτες που τη χρειάζονται. Ε, την τελευταία περίοδο βεβαίως έχει αυξηθεί η βοήθεια και μέσα από την Επιτροπή και διμερεί ε, προγράμματα κατορθώσαμε να επιτύχουμε περισσότερα από όσα είχαν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν βέβαια τεράστιες ανάγκες, η ε, διάθεση των προϊόντων είναι όλο και πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη και δυστυχώς δεν είναι εύκολη. Αυτά οφείλονται σε ένα διεθνές πλαίσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προαχθεί μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία όπου θα βασιζόμαστε στην ανεξαρτησία, την αμεροληψία, στην βοήθεια που θα πρέπει να φτάνει άμεσα και με αποτελεσματικότητα στα θύματα μιας κρίσης και ε, η βοήθεια θα δείτε με βάση τις ατομικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ένα λεπτό. Ο κύριος Αντωνιώτση. Οι φυσικέ καταστροφέ αυξάνονται τόσο αριθμητικά όσο και όσον αφορά την έντασή τους. Ε, πολλαπλασιάζονται οι κρίσει, και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιδείνωση της ε, παραβίασης ε, του ανθρωπιστικού δικαίου. Οι τελευταίες ε, τραγωδίες ε, στην Αϊτή και στο Πακιστάν καταδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν οι φυσικές ε, καταστροφές. Συμφωνώ λοιπόν με την γενικότερη θέση που ακολουθεί η έκθεση και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προάγει τις ανθρωπιστικές αρχές και μάλιστα ακούραστα. πρόκειται για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι λοιπόν απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ρίξει όλο τη το βάρο, ε, γιατί είναι οι βασικότερε φορέ που προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Αναφέρομαι στην έκθεση τη κυρία Στρίφλερ γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να θελήσουμε να δεσμευτούμε περισσότερο, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να προσφέρονται εγγυήσει για συντονισμό κυρίω ε, σε, παγκόσμιο επίπεδο και παράλληλα πρέπει να έχουμε κατά νου τις περιφερειακές ευθύνε που φέρουμε. Υπάρχουν χώρε που μπορούν να προσφέρουν περισσότερο περισσότερο στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστώ κύριε Αντωνιώτση. Και τώρα ο κύριος Χάναν για ένα λεπτό. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Χάναν. Τώρα όμως. Α, καλά. Δεν θέλετε. Ε, προχωρούμε. Στην έκθεση κυρία Σάρμπου. Γεωργία ο στρατηγικό τομέας στο πλαίσιο τη επιστημιστική ασφάλεια. Για ένα λεπτό, ο κύριο Χίγκεν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί επιβεβαιώνει ότι η ψηφιστική ασφάλεια είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ο γεωργικό τομέας θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του πληθυσμού που αυξάνονται για υγιεινά τρόφιμα. Παρόλο που είναι περιορισμένη η φυσική πόρη, ακριβή ενέργεια και έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με το ΦΑΟ, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 70% για να αντιμετωπίσουμε ε, τα 9 δισεκατομμύρια ε, πολιτών που θα έχουμε στον κόσμο το 2050. 900 εκατομμύρια ε, είναι χρονίως πεινασμένοι, υποσυτιζόμενοι λόγω της ένδυας και σε διάφορο βαθμό στην Ευρώπη 16% του πληθυσμού ε, ε, διαβεί κάτω του επίπεδου της φτώχειας. Τι εννοώ, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η χρηματοδότηση της νέας ΚΑΠ μετά το 2013 θα πρέπει να αναγνωρίζει ε, αυτή την ανάγκη. Και τουλάχιστον αυτό που χρειαζόμαστε είναι να διατηρηθεί ο προπολογισμό στα σημερινά του επίπεδα. Ευχαριστώ κύριε Χίγκενς και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Ρόντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε, αναγνώρισε σήμερα τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της επιστημιστικής ασφάλειας. Κάτι που ζητούσαμε εδώ και χρόνια. Επίσης αναγνωρίσαμε ότι η οικολογική γεωργία έχει στρατηγική σημασία για τη δημόσια υγεία και για την αηφόρο ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν τα σχολικά προγράμματα για τα τρόφιμα και το γάλα ή άλλα προγράμματα υποστήριξης ε, ε, του γάλακτος στα σχολεία είναι θετικά, γιατί με τέτοιες προτάσεις ε, μερικές φορές καταψηφίζονται. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε πρόθεση της γεωργίας, όχι όμως με τέτοια προγράμματα ένταξης του γάλακτος στα σχολεία, για παράδειγμα. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία ε, εξερεύνηση και νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας. Πάντως γενικώ η έκθεση είναι καλή, γι' αυτό και την υπερψηφίσαμε. Για ένα λεπτό το λόγο ο κύριος Μαστέλα. Πρόεδρε, η επιστημιστική ασφάλεια είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και αυτό πρέπει να ελοπιθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Μόνο όταν όλοι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, θα έχουν πρόσβαση φυσική, κοινωνική και οικονομική σε μια αποτελεσματική διατροφή, ε, μόνο τότε το ε, δικαίωμα αυτό θα έχει ε, γίνει σεβαστό. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με σαφή και διαμφισβήτητο τρόπο στις προκλήσεις που υπάρχουν, ε, κυρίως ε, να ανταπεξέλθουμε στην κλιματική αλλαγή, στην οικονομική κρίση, στην διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε να προάγουμε όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας, αλλά και την παραδοσιακή γεωργία, την κτηνοτροφία, την διανομή των προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. Αυτή λοιπόν η γεωργία ανέκαθε δεν ε, μας έδινε την επισητιστική ασφάλεια γιατί αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εδάφη σε συγκεκριμένε ε, περιοχές της ε, Ευρώπης και μέσα από μεθόδους οι οποίες έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένα για συγκεκριμένες περιοχές και για συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Στέλλα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ. Ο ρόλος μας ως Ευρωβουλευτών είναι να βελτιώσουμε, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα η εξασφάλιση της επιστηστικής ασφάλειας και ποιοτικών τροφίμων είναι ύψητη προτεραιότητα. Γιατί πολλές φορές οι πολίτες ανησυχούν για την εκτείναξη των τιμών των τροφίμων στα ύψη, για την έλλειψη ασφάλειας. Έχουμε τα προβλήματα τη δημογραφική ανάπτυξη, έχουμε πολλέ θεομηνίε, κλιματικέ αλλαγέ, γι' αυτό και η επιστηστική ασφάλεια ε, υπόκειται σε σημαντική απειλή. Και αυτό ανησυχεί τον κόσμο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και η οικονομική υποστήριξη του κλάδου τη γεωργίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα εκτακτό καθεστώ για τους ε, γεωργού για να ανταπεξέλθουν στην, στο ειδικό τους ε, λειτουργήμα και να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε η συμβολή του στις επιστημιστικές κρίσεις. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο ο κύριος Πυρίλο. Κύριε Πρόεδρε, η επιστημιστική ασφάλεια των πολιτών ε, αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση για τη Γεωργία, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή, αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο ε, για αυτά που ελαμβάνει η έκθεση, κυρίω διότι αναγνωρίζει ε, την ε, βοήθεια, την ασφάλεια αυτή ω ένα θεμελιώδη δικαίωμα των πολιτών. Ο στόχο τη επιστημιστική ασφάλεια, ο στόχο που είναι επιτευχθεί μόνο αν αντιμετωπίσει κανεί σοβαρά δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, τι διακυμάνσει τη αγορά και των τιμών και δεύτερον ε, το το περατό των πόρων. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση πρέπει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις στην επιστημιστική βοήθεια, να αντιμετωπίσει την ασυμμετρία που εξακολουθεί να υπάρχει όσον αφορά τα, τους όρους ε, της βοήθειας ε, που χορηγείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πυρίλο. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαπιστώσω ότι στην έκθεση αυτή χάρηκα πάρα πολύ ε, γιατί καταλαβαίνουμε και πάλι ποια είναι η σημασία της γεωργίας και τη φέρνουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας. Και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Σε ένα σημείο όμως ε, ψήφισα διαφορετικά και αυτό αφορά τη δημιουργία ενός ε, επισητιστικού προγράμματος βοήθεια στο εσωτερικό Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ νομίζω ότι επιτόπου βοήθεια, δηλαδή να μην επιτρέπεται κανείς να πεινάει στην Ευρώπη, αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει η αρμοδιότητα των κρατών μελών. Απλούστατα διότι ε, τα προβλήματα θα πρέπει να λύνονται εκεί που ε, εμφανίζονται και γεννιόνται, δηλαδή στα ίδια τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιά. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό η κυρία Ντότς. Η έκθεση αυτή τονίζει την ανάγκη επιστημιστική ασφάλειας και για τους πολίτες που εγώ εκπροσωπώ, αλλά τονίζει και τη ε, σημασία ε, των ε, αγαθών που παράγουν οι αγρότες με μικρή ή καμία αναγνώριση για τη δουλειά τους. Έχω ακούσει μεγαλόστομε δηλώσει πρόσφατα που δείχνουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα καταντήσει κοινή περιβαλλοντική πολιτική. Αυτό είναι λάθος. Γιατί τελικά μπορεί να εισάγουμε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε εκεί. Θα πρέπει να υποστηρίζουμε τους αγρότες για να παράγουν τρόφιμα με τρόπο ε, που δεν βλάπτει τον περιβάλλον. Και σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές τροφίμων, οι παγκόσμιες αγορές είναι πάρα πολύ πτητικές, πάρα πολύ ασταθείς και ως προς τις τιμές και ως προς την εξασφάλιση των εφοδιασμού. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε πολύ γερό προπολογισμό για την κοινή ευρωπαϊκή ε, πολιτική, την ΚΑΠ, ε, να έχουμε μέλλον για τους νέους αγρότες, περισσότερη έρευνα, περισσότερη καινοτομία, έτσι ώστε οι μέθοδοι παραγωγής να είναι πιο αποτελεσματικές, να μειώσουμε την γραφειοκρατία και κυρίως την γραφειοκρατία που έχει σχέση πλέον με το περιβάλλον, την οικολογία. Ευχαριστώ κυρία Ντότς. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Οζίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τις τελευταίες εβδομάδες οι διάφορες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής ασχολούνται με αυτό το θέμα, το θέμα της μεταρρυθμίσης που θα έχουμε από το, μετά το 2013. Τα βασικά στοιχεία της γεωργίας είναι σαφή. Ψηφιστική ασφάλεια είναι καθοριστικός παράγων. Έτσι λοιπόν το ε, πρέπει να εξελογηθεί σωστά και να έχουμε κατά νου ε, τις ε, διατάξεις που ψηφίσαμε σήμερα. Η ασφάλεια αυτή είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ως τέτοιο θα πρέπει να προστατεύεται με όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Βεβαίως, Πρόεδρε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και κάποιες έκτακτες συνθήκες όπως το σκάνδαλο με τις διοξίνες, ένα σκάνδαλο που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες και αφορά στην ζώων. Αλλά να έχουμε κατά νου και τις ε, καθημερινές δραστηριότητες ε, που αφορούν στην ε, παραγωγή των προϊόντων. Να έχουμε κατά νου την ποιότητα αλλά και την προστασία των καταναλωτών. Πρόκειται λοιπόν για μια διάταξη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μαζί με άλλε επίση διατάξει που αφορούν στην κοινή γεωργική πολιτική. Εγώ λοιπόν δηλώνω ότι είμαι ευχαριστημένο με αυτέ τι δραστηριότητε. Σα ευχαριστώ για ένα λεπτό τώρα ο κύριο Μετσάρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παραγωγή τροφίμων στον κόσμο είναι εκτεθειμένη σε όλο και περισσότερες απειλές. Μία απειλή είναι οι κλιματικές αλλαγές, που είναι και απρόβλεπτες και μπορεί να θέσουν σε ισχύ την, ε, τον ανεφοδιασμό τροφίμων 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, που θα είναι ο πληθυσμός της γης το 2050. Η κοινή γεωρική πολιτική θα πρέπει να δώσει απάντηση στις προκλήσεις της επιστημιστικής ασφάλειας, όχι μόνο ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, αλλά υποστηρίζοντας και την παραδοσιακή γεωργία, τα μικρά αγροκτήματα και τους τοπικούς συνεταιρισμούς. Εξαιτία των κλιματικών αλλαγών έχουμε όλο και περισσότερες θεομηνίες και φυσικές καταστροφές που πλήττουν τη γεωργία και δεν επιτρέπουν αποτελεσματική χρήση μεγάλων εδαφικών εκτάσεων. Θα πρέπει παρόλα αυτά να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπέ εισόδημα στου γεωργού. Γι' αυτό και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και με τον προπολογισμό την κοινή γεωργική πολιτική. Η γεωργία θα πρέπει να θεωρηθεί ω στρατηγικό τομέα σε θέματα επιστημιστική ασφάλεια, γι' αυτό και υπερψηφίσαμε τη σχετική έκθεση. Σα ευχαριστούμε κύριε Ματσάρο. Για ένα λεπτό, το λόγο έχει ο κύριο Ταραμπέλα. Απουσιάζει ο κύριο Ταραμπέλα, οπότε για ένα λεπτό το λόγο ο Στάκουλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναγνώριση της σπουδαιότητας της Γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισητιστικής ασφάλειας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα τρόφιμα που παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ποιοτικά, υγιεινά και οικολογικά. Με ανησυχεί ότι δίνουμε περισσότερη έμφαση στην ποσότητα από ό,τι στην ποιότητα. Φαίνεται ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο η αποτελεσματικότητα από το χαρακτήρα, το υγιεινό χαρακτήρα των τροφίμων. Οι καταναλωτές όμως ενδιαφέρονται για ποιοτικά τρόφιμα, για υγιεινά τρόφιμα που θα βρίθουν θρεπτικό συστατικών. Αυτό θέλει ο καταναλωτής. Θα πρέπει λοιπόν να παράγουμε τρόφιμα που θα παράγονται με παραδοσιακούς γεωργικούς τρόπους για να εξασφαλίσουμε και μια αυτάρκεια και έναν επισητιστικό ανεφοδιασμό και να παράγουμε κυρίως τρόφιμα ντόπια για να αποφύγουμε και τι επιστημικές κρίσει. Η υγεία φυσικά είναι σοβαρότατο παράγοντα. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα τα τρόφιμα να είναι υγιεινά και να παράγονται, όπω είπα, όλο και περισσότερο σε τοπικό επίπεδο τα τρόφιμα. Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά ε, και τα, και τα κράτη-μέλη μπορούν να, συνεχίσουν να τροφοδοτούν ε, την τοπική τους γεωργία. Νομίζω ότι θα είναι σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Ο κύριος Σταταρέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ε, έχοντας ε, πει ότι είμαι υπέρ αυτής της ε, έκθεσης. Εκείνο που θέλω είναι να υπογραμμίσω ιδιαίτερα το σημείο υπαριθμών 35 της έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, όπου αναφέρεται η σημασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την επισητιστική ασφάλεια. Είναι σημαντική αυτή γιατί μπορεί να αξιολογήσει όλους τους κινδύνους που υπάρχουν στον επισητιστικό κλάδο ε, και είναι σημαντικό να προστατεύεται ο πολίτης και η υγεία. Εκφράζεται επιπλέον η ευχή όλα τα κράτη-μέλη να ε, προσφέρουν στον οργανισμό αυτό την συνεργασία με τους εθνικούς τους οργανισμούς γιατί ε, όπως σα είπα, ο απότερο στόχο είναι η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Στη Γερμανία είχαμε πρόσφατα εξελίξει και αυτές καταδεικνύουν κάθε κράτο να έχει το δικό του τον οργανισμό για την επισητιστική ασφάλεια. Η Ιταλική κυβέρνηση έχει συστήσει έναν οργανισμό, μετά όμω δυστυχώ άλλαξε γνώμη και αυτό για δημοσιονομικού λόγου. Εγώ όμω θεωρώ ότι η επισητιστική ασφάλεια δεν θα πρέπει να παραβλέπεται λόγω δημοσιονομικών δυσκολιών. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνονται λοιπόν εδώ η επεξηγήση ψήφου. Διακόπτεται η συνεδρίαση έως τις 3. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι.